ελληνικές αρχές με ενημέρωσαν πως η ποινική διαδικασία κατά του κυρίου Σωτηρίου Ζαριανόπουλου για την οποία είχε αρθεί η ασυλία του έχει πλέον ολοκληρωθεί και μπει στο αρχείο.